θα σας ε, δημοσιευθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Την ε, Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συνομπουλίου, θα υπογράψω δύο ε, νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία. Τους τίτλους θα τους βρείτε επίσης στα πρακτικά της συνεδρίασης. Για το κανονισμό, για το δικαστικό ζήτημα μάλλον, το λόγο ζητάει ο κύριος Κάρθη. Έχει το λόγο. Mr. μετά την τελευταία μας συνάντηση στο στην Ιρλανδία αντιμετωπίσαμε ε, μια τρομερή καταστροφή. Δέκα μέλη της ε, κοινότητας των ταξιδιωτών, των ομάδων στην Ιρλανδία έχασαν τη ζωή τους. Θα ήθελα να στείλουμε στις οικογένειές τους τα συλληπιτήρια του Κοινοβουλίου επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Τόνι Γκόλνταν, μέλος της ειρηνευτικής, ε, του ειρηνευτικού τμήματος του στρατού της Ιρλανδίας, ε, έχασε τη ζωή του και θα ήθελα και σε αυτή την περίπτωση να στέλνουν συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θα ελέγξουμε τη διαδικασία, κύριε Κάρτη, εννοείται, και θα πράξουμε ένα για το διαδικαστικό ζήτημα Λοιπόν, βάσει του άρθρου ε, 286, το λόγο Ζήτησε ο κ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε μια κατάσταση που εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρή και έχει σχέση με μια παράλογη επέμβαση των υπηρεσιών των οποίων υγείστε εσείς με τις παρεμβάσεις στις, ε, ε, στους χρόνους αγόρευσης των ε, Ευρωβουλευτών. Ευρωβουλευτών, υποχρεώνοντας σε γραπτές απαντήσεις και σε νέες εκτιμήσεις ε, της Κομισιόν όσον αφορά την Επιτροπή ε, των Συνταγματικών Υποθέσεων. Οι αιτιολογήσεις ψήφους αλλά και οι αιτιολογήσεις για τα κατεπήγοντα αμφισβητώνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις και επί ποιας βάσεως. Επί ποιας βάσεως αποφασίζεται αν είναι θεμητή ή όχι η αιτολόγηση ενός κατεπήγοντος ζητήματος που υποβάλλει ένας βουλευτής. Ε, θέλω να γνωρίζω, θέλουμε να γνωρίζουμε ποιος λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις και επί τη βάση ποιων αρχών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ζωάφερα. Με ενημερώνουν οι υπηρεσίες μας ε, ότι θέλετε να θέσετε το θέμα αυτό και στην παρούσα φάση πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ να σας παρουσιάσω την ερμηνεία του άρθρου 130, αλλά μετά από ανάλυση του αιτήματό σας, μόλις ολοκληρωθεί μάλλον η ανάλυση αυτή, θα σας ε, διαβιβάσουμε άμεσα τα πορίσματα. Κυρίε και κύριοι, από τη διάσκεψη του Προέδρου βάσει του άρθρου 149 ε, στις 22 Οκτωβρίου ε, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη και σας προτείνω εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων να γίνουν εξής αλλαγές στην τελική ημερήσια διάταξη. Οι δύο δηλώσεις της ε, Αντιπροέδρου της